Good um, Ο Πρόεδρος. Καλή σας μέρα, συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στα έδρανά σας και ελπίζω να περάσετε καλές θερινές διακοπές. Σας αρχίσουμε με την έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Αν δεν έχετε ενστάσεις, τότε θεωρώ ότι εγκρίνεται. Πρώτα, για το γλωσσικό καθεστώς έχουμε τις διάφορες γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Ας αρχίσουμε πρώτα με την έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Ο κύριος Βύση του ECR ορίστηκε συντονιστής για θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Ο κύριος Διαστεμέρα του Λαϊκού Κόμματος για την απόφαση του Συμβουλίου για το κεκτημένο Σέγγεν, για το σύστημα πληροφοριών προξενικών θεωρήσεων. Ο κύριος Ντάλτον του ECR εισηγητής για το EQUIS. Παρακαλώ πολύ ησυχάστε για να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Η κυρία Σαρτζεντίνη ορίστηκε η συγγήτρια για την ε, κατάσταση στην Ουγγαρία, πρόταση νομοθετικού περιεχομένου που υποβλήθηκε στις 17 ε, Μαΐου 2017. Ο κύριος Κρυπέκ από το ECR ε, ασχολείται με θέματα διαλειτουργικότητας για τα οδικά δίκτυα. Αυτά. Εγκρίνονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε ορισμένες πληροφορίες για τις κατεξιοδότηση πράξης. Στις 24 Αυγούστου 2017 εγκρίθηκε το πρόγραμμα για τις δράσεις στα πλαίσια του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί το έγκλημα και η διαχείριση κρίσεων. Η βασική νομοθετική πράξη Ευρωπαϊκή Ένωση 514-2014 είναι η βάση. Με βάση τη διαδικασία επιτροπολογίας και υπάρχει και η προθεσμία προτάσεων. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις, παρακαλώ να ενημερώσετε τη Γραμματεία ΛΥΜΠΕ πριν από τις 8 Σεπτεμβρίου 10. Και επίσης στις 11 έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, γι' αυτό σας παρακαλώ να έχετε έτοιμες ε, τις κάρτες σας. Στη συνέχεια έχουμε την έγκριση των παρακτικών ε, της 9ης και 27ης Μαρτίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά. Άρα φτάνουμε στο σημείο 4 που είναι η πρόσφατη εξελίξη στην Πολωνία και ο αντίκτυπο του στο κράτος δικαίου. Θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων τον, με τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Φραν Τίμερμανς. Σε καλωσορίζουμε Φρανς και πριν ε, λάβει το λόγο, ας μιλήσουμε για τα γεγονότα. Στις 26 Ιουλίου 17 η Επιτροπή ενέκρινε μία σύσταση σε σχέση με το κράτος δικαίου στην Πολωνία με βάση δύο συστάσεις του 16. Όπως γνωρίζετε, στις 13 Ιανουαρίου 2016 η Επιτροπή ξεκίνησε έναν διάλογο για την κατάσταση στην Πολωνία με βάση το πλαίσιο για το κράτος δικαίου και επειδή υπάρχει, ε, υπάρχουν νομικές διαφορές σε σχέση με τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και την ε, μη ε, έκδοση των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου καθώς και την αναθεώρηση του συνταγματικού δικαίου στη, κατά την, την 1η Ιουνίου 2016 η Επιτροπή ενέκρινε τη γνωμοδότηση για την κατάσταση δικαίου στην, στην Πολωνία και αυτό με βάση τις ε, ε συστάσεις της 27ης Ιουλίου και 21ης Δεκεμβρίου ε, 16. Όπως ξέρετε οι συστάσεις ε, παρουσιάζουν το όλο σύστημα με πολλές ανησυχίες σε σχέση με τον διαχωρισμό των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Γι' αυτό οι πολωνικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν κατεπηγόντως το θέμα της διατάραξης του κράτους δικαίου. Η σύσταση της Επιτροπής ζήτησε από τις πολωνικές αρχές να αντιμετωπίσουν το ζήτημα μέσα σε ένα μήνα. Σήμερα στην Επιτροπή μας θα θέλαμε να ακούσουμε καταρχήν τον πρώτο αντιπρόεδρο Φρανς Τίμερμανς και να προβούμε σε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα ακούσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο και στη συνέχεια θα προβούμε σε ανταλλαγή ε, απόψεων δυνάμει του άρθρου 206 καταρχήν θα λάβουν το λόγο μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και στη συνέχεια βουλευτές από άλλες επιτροπές. Ο κύριος Τίμερμανς θα λάβει το λόγο για 10 λεπτά. Θα ήθελα να ε, αναφέρετε κατά πόσο θέλετε το λόγο. Καταρχήν οι συντονιστές, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και τα υπόλοιπα μέλη. Το λόγο έχει ο πρώτος αντιπρόεδρος και στο τέλος θα απαντήσει τις ερωτήσεις. Έχουμε μια μισή ε, ώρα, φαίνεται πολύ, όμως δεν είναι πολύ η ώρα. Έχετε, ε, μπορείτε να λάβετε το λόγο για δύο λεπτά, θα χρονομετρηθείτε και θα ήθελα να αρκεστείτε στα ε, δύο λεπτά. Και η γραμματεία θα καταγράψει τα ονόματά σας. Φρανς, Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Την περασμένη φορά που μιλήσαμε για αυτό το θέμα στην Επιτροπή αυτή ήταν στις 22 Μαρτίου και σήμερα έχω το καθήκον να σας ενημερώσω για τα όσα έχουν συμβεί από τότε. Τέσσερις νόμοι έχουν υιοθετηθεί από το Πολωνικό Κοινοβούλιο από τότε. Ε, για το δικαστικό σύστημα, την διοίκηση και την οργάνωση των δικαστηρίων, για το ανώτατο δικαστήριο και το Εθνικό Συμβούλιο, ε, το δικονομικό. Στα τέλη Ιουλίου, μετά από εντελεχή ανάλυση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα τέσσερα αυτά νομοσχέδια, οι τέσσερι νόμοι που έχουν υιοθετηθεί, θα έχουν ένα πολύ αρνητικό αντίκτυπο ε, στην ανεξαρτησία τη ε, πολωνική δικαιοσύνη και θα αυξήσουν το συστημικό κίνδυνο και την απειλή για το κράτο δικαίου αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ε, έχει ε, τεθεί η δικαίωμα κυρίας για τους δύο από τους τέσσερις νόμους από τον πρόεδρο Τούδα, όμως το γεγονός ότι δύο από τους τέσσερις νόμους έχουν ε, υπογραφεί σημαίνει ότι θα πρέπει πραγματικά να μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα ε, σε μια νέα σύσταση για το κράτο δικαίου. Η τρίτη σύσταση που απευθύνθηκε στην Πολωνία στι 26 Ιουλίου συμπληρώνει τι προηγούμενε, και παρουσιάζει τι σοβαρέ ανησυχίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, προτινόμενες αλλαγέ ε, του δικαστικού συστήματο στην Πολωνία. Επίση, ζητά από τι πολωνικές αρχέ να αποκαταστήσουν την ανεξαρτησία και την νομιμότητα του συνταγματικού δικαστηρίου ως θέματοφύλακα του πολωνικού Συντάγματο. Ζητούμε λοιπόν οι πολωνικές αρχές να εξετάσουν αυτές ε, τις παρατηρήσεις εντός ενός μηνός. Στις 28 Ιουλίου επίσης η ε, Επιτροπή Κίνηση δικασία Επιπαραβάση κατά της Πολωνίας για την παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου ε, για την οργάνωση και διοίκηση των τακτικών δικαστηρίων και επίσης ζητήσαμε να δοθεί απάντηση εντός του μήνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πάνω από ένα χρόνο παρουσίασε τις Παρατηρήσει τη για την κατάσταση του κράτου δικαίου στην Πολωνία. Έχουμε αναλύσει, έχουμε εντοπίσει ζητήματα, έχουμε προειδοποιήσει, έχουμε στείλει τρεις συστάσεις, έχουμε κινήσει διαδικασία επί ε, κατά τη Πολωνία. Για να συμπληρώσω αυτή την ε, επισκόπηση, να γνωρίζετε ότι δεν αρνείται η πολιτική κυβέρνηση να ακολουθήσει τα ενδιάμεσα μέσα μέτρα που έχει υιοθετήσει ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για συγκεκριμένους τομείς, για τα δάση, αλλά και για την αποκέντρωση των ε, μέσων ενημέρωσης, όπως αναφέρεται. Και ο πρόεδρος απέστειλε επιστολή στις αλβανικές αρχές, όπου παρουσιάζονται οι ε, παρατηρήσεις ό,τι αφορά τις ε, διαφορές στην ηλικία σταξιοδότησης ανδρών και γυναικών. Η Πολωνία αυτή τη στιγμή είναι μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που πλέον είναι ε, κινδυνεύει να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση σχέση με τι υπόλοιπε. Στις 28 Αυγούστου λάβαμε απάντηση στην τρίτη σύσταση. Πριν την απάντηση, η πολωνική κυβέρνηση δύο φορές ε, ζήτησε περισσότερε διευκρινήσει για τους δικού μα προβληματισμού που εμείς ε, αμέσως και πολύ εντελεχώ στείλαμε. Ακόμα αναλύουμε με μεγάλη προσοχή την απάντηση. Όμως και από Δηλώσει των βαλικών αρχών μπορώ να σα πω ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο μέτρο που να προκύπτει από την πολωνική απάντηση που θα καλύπτει και θα διασκεδάσει τις ανησυχίε μα. Εμεί θα επικεντρωθούμε πολύ συγκεκριμένα ε, στις ε, αιτιολογήσει που μα έχουν δώσει αλλά δεν μπορώ να σα πω σήμερα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τη Επιτροπή. Θα πρέπει να το εξετάσω και με το Σώμα των Επιτρόπων και κάποια στιγμή θα ε, το υποβάλουμε και στο Συμβούλιο. Ωστόσο να κάνω κάποιε γενικέ παρατηρήσει. Έχουμε αφιερώσει μεγάλη μεγάλο χρόνο και ενέργεια και πολλές σελίδες ε, στην παρουσίαση αυτών των ε, απαντήσεων και το κάναμε όσο μπορούσαμε πιο εντελεχώς. Επίσης ε, υπάρχει ευρεία συνένεση ότι αφορά αυτές τις παρατηρήσεις από την Επιτροπή της Βενετίας, τον ΟΗΕ, το Δίκτυο των Δικαστηρίων, Ενώσεις Δικηγόρων και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Στις 16 Μαΐου είχαμε μια πρώτη εκτενή ε, συζήτηση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και υπήρξε ε, ευρύτατη συμφωνία ότι το κράτος δικαίου είναι κοινό συμφέρον και κοινή αρμοδιότητα των ευρωπαϊκών θεσμών και κρατών μελών. Η ε, ευρύ πλειοψηφία των κρατών μελών στηρίζει τις προτάσεις και τις ε, τις προτάσεις αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλουμε να επιλύσουμε τα εκκρεμή ζητήματα και αναμένουμε να ενημερωθούμε ε, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Περιμένουν τα κράτη-μέλη μάλλον να ενημερωθούν. Έχουμε καλέσει και του ε, Πολωνού Υπουργού να έρθουν στι Βρυξέλλε για να τα συζητήσουν αυτά τα θέματα μαζί μου. Δεν έχω λάβει ακόμα ε, επίσημη απάντηση, αλλά στα μέσα ενημέρωση ε, είδαμε ότι υπάρχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο, δεν βρίσκουν κάποιο λόγο να έρθουν και να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Εμεί βέβαια θα το θέλαμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, οπότε όποτε θελήσουν ε, να έρθουν, εμείς ε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα προφανώς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και τώρα και στο μέλλον. Είναι άμεσα εκλεγμένο και το βασικό καθήκον αυτού του Κοινοβουλίου είναι η υπεράσπιση των κοινών ευρωπαϊκών μα ε, αξιών. Και το κράτο δικαίου είναι ε, ακρογωνιαίο λήθο αυτό. Η πολωνική κυβέρνηση επανειλημμένω έχει δείξει ότι δεν αποδέχεται αυτέ τι παρατηρήσει Επίσης, ε, στρέφεται κατά ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απλώς μεταφέρει την κατάσταση και αναφέρει το προφανές και λέει ότι δεν κάνει τίποτα διαφορετικό από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Εγώ προσωπικά διαφωνώ. Πάντα λέμε ότι ο στόχος μας δεν είναι η επιβολή κυρώσεων ε, η επίκληση του άρθρου 7. Αντιθέτω, θέλουμε έναν πραγματικό ε, επικαθηματικό διάλογο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του κράτου δικαίου στην Πολωνία. Ωστόσο, έχουμε επίση ξεκαθαρίσει ε, ότι είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα ω θεματοφύλακε των συνθήκων, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Και παραμένουμε ανοιχτοί στο διάλογο και στην εξέβρεση επικαθηματικών λύσεων. Ταυτόχρονα όμω πρέπει να συζητήσουμε και εσωτερικά στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο με τα κρατημέλη και με εσά εδώ στο Κοινοβούλιο τη νέα κατάσταση όπω έχει διαμορφωθεί. Εμεί δεν το αφήνουμε, δεν κάνουμε πίσω και αυτό έχει να κάνει με δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, προφανώ το κράτο δικαίου από μόνο του έχει πολύ μεγάλη αξία. Είναι η ταυτότητά μα. Είναι αυτό που μα προσδιορίζει ω Ευρωπαίου πολίτε μία δημοκρατία βάσει του κράτους δικαίου. Δεύτερον, έχει να κάνει και με τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα η ενιαία αγορά. Αυτή η αγορά μπορεί μόνο να λειτουργήσει αν υπάρχει ε, πραγματική εμπιστοσύνη μεταξύ κυβερνήσεων, εμπορευομένων, οικονομικών φορέων, ε, πολιτών που πραγματικά πιστεύουν και είναι σίγουροι ότι όπου υπάρχει ε, κάποια ε, νομική διαφορά ε, όλοι είμαστε ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουμε πρόσβαση σε ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα. Και οι εθνικοί δικαστές, οι δικαστές των κρατών μελών είναι και ευρωπαίοι δικαστές γιατί εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και έχουν και απρόσκοπτη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και αυτό δεν μπορεί να σταματήσει γιατί υπάρχει ε, πολιτική παρεμβολή και παρέμβαση των κυβερνήσεων. Η ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματο είναι θεμελιώδη σημασία για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού συστήματο. Πρέπει ε, να είμαστε σίγουροι ότι οι δικαστέ των κρατών μελών είναι και Ευρωπαίοι δικαστέ. Ιδάλλως, εάν επανέλθουμε σε μια κατάσταση όπου το κράτος δικαίου εξαρτάται από ένα τηλεφώνημα που θα κάνει ένας πολιτικός ε, σε μια χώρα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Οπότε η ανεξαρτησία των εθνικών δικαστών είναι βασικό στοιχείο για τη συνεργασία των ε, κρατών μελών ε, στον ε, τομέα της δικαιοσύνης και των ιστορικών υποθέσεων. πρέπει να μιλήσουμε και για την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και ο κανονισμός Βρυξέλλες 1. Βεβαίως, δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις σαφώς και έχουν το ελεύθερο να ε, υιοθετήσουν και να υλοποιήσουν δικαστικέ μεταρρυθμίσει. Εμεί δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα τη πολιτική κυβέρνηση να ε, προβεί σε δικαστική μεταρρύθμιση καθόλου. Όμω, ισχυριζόμαστε ότι η δικαστική μεταρρύθμιση θα πρέπει να τηρεί το κράτο δικαίου. Ω ε, μία από τι βασικές αρχές που έχουν προσυπογράψει όλες ε, οι χώρες, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν ε, εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπέγραψαν τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Όποιο ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να μην υπάρχει παρέμβαση πολιτικών και άλλων φορέων. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις για όλα αυτά. Η τήρηση και η περάσπιση του κράτους δικαίου είναι κοινή αρμοδιότητα και ευθύνη όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ε, έχω κάθε πρόθεση βέβαια να συζητήσω αυτό το θέμα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, όπως συμφωνήσαμε το Μάιο, και θα τους ενημερώσω. Εν κατακλείδη θα ήθελα να ευχαριστήσω εσά και πιο συγκεκριμένα την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για τι συνεχεί προσπάθειε για την υπεράσπιση του κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη στήριξη που έχετε απευθύνει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την κατάσταση στην Πολωνία. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρο, σας ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ κύριε Πρώτε Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ και για την συντομία του λόγου σας. Βεβαίω τώρα όλα τα παρόντα μέλη επιθυμούν να λάβουν το λόγο και αυτό είναι κατανοητό. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να ασκήσετε πειθαρχία και να είστε συνεκτικοί. Όλα τα παρόντα μέλη είναι εγγεγραμμένα, που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να υπερβείτε τα δύο λεπτά. Πάντως, θα παρακαλέσω και τους συντονιστές και συντονίστριες να αρκεστούν στα δύο λεπτά και μετά να ακούσουμε, μετά από τους συντονιστές δηλαδή, μια πρώτη σύντομη απάντηση από τον κύριο πρώτο αντιπρόεδρο. Όλοι όσοι έχουν δηλώσει ως τώρα ότι επιθυμούν να λάβουν το λόγο είναι εγγεγραμμένοι. Και τώρα κλείνω τον κατάλογο. Αρχίζω πρώτα με την κυρία Μεζόλα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς κύριε αντιπρόεδρε. Υπογραμμίζω ότι η κατάσταση στην Πολωνία μας ανησυχεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε το θέμα του κράτους δικαίου στην χώρα αυτή και υποψιάζομαι ότι θα είναι και η τελευταία. Μεγάλωσα στην ε, Μάλτα παρακολουθώντας ε, τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Δεύτερο και την Solidarność ε, στην Πολωνία που πρόσφεραν ελπίδα στον κόσμο. Ελπίζω ότι η δικαιοσύνη εν τέλει θα κατησχύσει. Βλέπουμε ότι ο πολωνικός λαός άναψε τότε μια φλόγα που ελπίζω η παρούσα γενεά να μην την δει ποτέ να σβήνει. Γι' αυτό και έχει ενταχθεί η χώρα αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι Πολωνή, όμως είμαι και Ευρωπαία. Έχουμε λοιπόν μια κοινή αγορά, έχουμε κοινά σύνορα και κυρίως έχουμε κοινέ αξίες. Η Ευρωπαϊκή μας Ένωση οφείλει να αρθεί στο ύψος των αξιών αυτών, να ταχθεί υπέρ της ανεξαρτήθειας δικαιοσύνης και στην Πολωνία και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και σωστά ενέκρινε τις συστάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Πολωνία. Σωστά έπραξε και υπερασπίζεται τις αξίες της και τις αξίες μας. Αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι να δράσει υπέρ θεμάτων όπως η δικαιοσύνη. Βλέπουμε την πλευρά της πολωνικής κυβέρνησης να προβάλλει τα ίδια επιχειρήματα ότι δήθεν η Ευρώπη ανακατεύεται εκεί που δεν πρέπει προβάλλοντας λαϊκίστικα επιχειρήματα και νομικά ασφαλμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να δράσει όταν απειλείται το κράτος δικαίου και σωστά έπραξε. Όμως οι απειλές κατά του κράτους δικαίου στην Πολωνία δεν έχουν ξεπεραστεί. Ο νόμος για το ανώτατο δικαστήριο και για το Ανώτατο Συμβούλιο μπορεί να αντιμετωπίστηκαν με βέτο από τον Πολωνό Πρόεδρο μετά από ημέρες διαμαρτυριών του κοινού. Γνωρίζουμε όμως ότι Τώρα προωθούνται νέα νομοσχέδια και δεν, δεν γνωρίζουμε ποια μορφή θα λάβουν. Άλλα δύο νομοθετήματα για τα ε, κοινά δικαστήρια και για την ε, δημοσίευση των αποφάσεων, γνωρίζω και τα σχόλιά σας κύριε Αντιπρόεδρε, ακολουθούν. Τι θα γίνει λοιπόν, ποιες είναι οι προσδοκίες σχετικά με το ότι οι πολωνικές αρχές θα απαντήσουν σε πνεύμα επικοδομητικής συνεργασίας Πρέπει να γίνει αυτό, διότι αλλιώ η εξέλιξη θα είναι αρνητική. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που έχετε οργανώσει την σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα να έλθω ιδίω σε ορισμένα σχόλια. Όλοι από τότε που ιδρύσαμε το την εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση βασιστήκαμε στην αρχή ότι είναι φυσικό ότι όλες οι χώρες μέλη μας είναι αυτονόητο ότι θα ακολουθούν τους κανόνες και τις αξίες τους κανονισμούς και τις ε, οδηγίες που έχουμε συναποφασίσει και ότι θα σέβονται τις αρχές και τις αξίες της συνθήκης. Τα θεωρήσαμε όλα αυτά αυτονόητα. Ίσως γι' αυτό οι δυνατότητες μας να αντιδράσουμε σε περιπτώσεις όπου αυτό δεν συμβαίνει είναι κάπως αδύναμες. Βλέπω ότι οι επικρίσεις δεν προέρχονται μόνο από το Κοινοβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από τους ίδιους τους Πολωνούς πολίτες. Και αυτό με ικανοποιεί. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως σε μια περίπτωση όπου μια χώρα μέλος δεν ακολουθεί τους κανόνες τους οποίους έχει συνυπογράψει. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαδικασία παραβιάσεως, επί παραβιάση. Αλλά αυτή η διαδικασία παίρνει πολύ χρόνο και τα πράγματα μπορούν να εξελίσσονται στο μεταξύ. Έχουμε και το άρθρο 7. Αλλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το άρθρο 7 θεωρούνταν ως κάτι υπερβολικά επικίνδυνο. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν τα χέρια μας είναι δεμένα και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε με ένα ευεξήγητο τρόπο. Εγώ υποστηρίζω πάντοτε ότι τα πρώτα βήματα θα πρέπει να είναι να δοθεί μια πολύ φιλική συμβουλή στη συγκεκριμένη κυβέρνηση εξηγώντας ότι έχουν λάβει μια οδό που ενδεχομένως να θέσει σε κίνδυνο τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Εάν δεν αντιδράσουν με τον τρόπο που αναμένουμε ωστόσο οι κυβερνώντες χρειάζεται να έχουμε και άλλους τρόπους και να εξοικονομήσουμε και χρόνο για τις αλλαγές αυτές, να μην περάσει πολύς χρόνος. Ο κύριος Γιούρεκ που αντικαθιστά την κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για τις ευρωπαϊκές αξίες. Εκπλήσωμε που δεν θυμήσατε ότι σήμερα είναι η 37η επέτειος της νίκης των Πολωνών εργατών των ναυπηγείων του Γκτάνσκ. Δεν είναι μονάχα πολωνική επέτειος αυτή, είναι και ευρωπαϊκή επέτειος, διότι οι Πολωνοί εργάτες άνοιξαν τον δρόμο προς την ελευθερία στην κεντρική Ευρώπη και την ασφάλεια για όλη την Ευρώπη. Θα συνεχίσω όμως μετά την γαλλική αυτή παρέμβαση στα πολωνικά. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, έχετε το δίκαιο, βεβαίως έχετε δίκαιο να έχετε διαφορετική άποψη. Αλλά η δράση που αναλαμβάνετε πρέπει να είναι σύνομη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να απευθύνει κατηγορίες σε οποιαδήποτε χώρα, είτε είναι η Πολωνία, είτε η Τσεχία, είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα, η Ουγγαρία κλπ, ότι παραβιάζουν κάποια άρθρα των συνθήκων. Πρέπει όμως να υποβάλει την αίτησή της αυτή στο Συμβούλιο Υπουργών και να αναμείνει υπομονητικά τη δική του απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να σεβαστεί το γεγονό ότι δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των χωρών μελών σε ό,τι αφορά τι καταγγελίε κατά της Πολωνία. Εγώ μίλησα για την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία επίση αξίζει τον σεβασμό μα Το ίδιο το πολωνικό σύνταγμα. Δεν μπορείτε να λέτε, για παράδειγμα, για τα δικαιώματα των γυναικών ή για την πρόορη συνταξιοδότηση. Δεν μπορείτε να λέτε ότι αυτά τα πράγματα αποτελούν διακριτική μεταχείριση και ταυτόχρονα να ζητείτε η διατήρηση του Συνταγματικού Συμβουλίου, διότι το ίδιο αυτό Συμβούλιο το 2010 είπε ότι το δικαίωμα πρόορης συνταξιοδότησης είναι δικαίωμα του καθενός και συνταγματικό δικαίωμα και των γυναικών. Έτσι λοιπόν σας παρακαλούμε να σεβαστείτε το σύνταγμά μας και να μην χρησιμοποιείτε τον νόμο ως εργαλείο. Διότι εμείς έχουμε ξεμπερδέψει πλέον με τον μαρξισμό, ο οποίος θεώρησε το δίκαιο και τον νόμο σαν εργαλείο για την επιβολή του. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γενικά γιατί οι συνάδελφοι θα μιλήσουν για την κατάσταση στην Πολωνία, θα μιλήσουν για τις ανησυχίες τους αλλά και τις ελπίδες τους από τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον κύριο Τίμερμανς, για την παρουσία του στην Επιτροπή μας ε, σήμερα το πρωί που αποδεικνύει την ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών, γιατί θα πρέπει να προωθήσουμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Τον ευχαριστώ γιατί μας υπενθύμησε και τις βάσεις αυτής ε, της ε, αποφασιστικότητας, γιατί είμαστε θεματοφύλακες των συνθήκων και θέλουμε πραγματικά να έχουμε να κάνουμε με μια συμμετοχική Ευρώπη με όλα τα κράτη εξασφαλίζοντας το συλλογικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, υπεράσπιση των αξιών μας. Κατά τις τελευταίες εβδομάδες ε, ξετυλίχθηκαν αυτές οι ανησυχίες, αλλά και ο διάλογος και η εργαλειοθήκη των συνθήκων ο συνάδελφος Μπρόνισλαφ Γκέρεμεκ θα είναι πολύ ανήσυχος και λυπημένος για το τι συμβαίνει σήμερα από τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την ε, πολωνική κυβέρνηση. Είναι σαν να προωθούμε μία διελκυστίνδα αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ε, εμείς δεν αμφισβητούμε τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και ευχαριστώ τον κύριο Τίμερμανς που το υπενθύμησε. Εμείς ε, δεν θέλουμε να κλιμακώσουμε μία αντιπαράθεση θέλουμε να προωθήσουμε μία γενικευμένη συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων πολιτών και να αμφισβητήσουμε ε, την ε, ε, αντιπαράθεση στη μνήμη του Μπρόμισλαφ Γκέραμεκ. Η κυρία Σπινέλη έχει το λόγο από τους συντονιστές. Ευχαριστώ πρόεδρε. εγκρίνω απόλυτα τις πρωτοβουλίες και συστάσεις της Επιτροπής και θα ήθελα να υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά ίσως μία παρεξήγηση σε σχέση με την φύση και την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το λέω γιατί είδα την αντίδραση τη Δευτέρα της πολωνικής κυβέρνησης στις συστάσεις της Επιτροπής. Η απάντηση αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προσδοκίες του λαού μέσα στα πλαίσια της πολωνικής ταυτότητας. Όμως η συνταγματική μας δημοκρατία ορίζει ως πρόκριμα για την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τήρηση των κανόνων του ε, κράτους δικαίου. Και εδώ δεν πρόκειται για μία αφηρημένη έννοια. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο όπου εντάσσονται και οι κοινωνικές προσδοκίες. Άρα αυτό αυτή η παρεξήγηση θα πρέπει να αποσαφινιστεί. Επίσης, και σε σχέση με αυτή την ε, παρεξήγηση θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο η Επιτροπή θα αποσαφηνίσει ε, τη θέση της σε σχέση με τις χώρες ε, της ομάδας του Βίζεγκραντ που θα συναντηθούν αύριο για μία νέα διάσκεψη τέλος το άρθρο 7 αρκεί ως αποτρεπτικό μέσον γιατί δυστυχώς ε, δεν υπάρχει πλειοψηφία κρατών για να ταχθεί πέρα αυτού και να κινήσει τη διαδικασία. Μιλήσαμε και για άλλα μέσα και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι αυτά για να αρθεί η παρούσα κατάσταση. Η κατάσταση αυτή αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο την Πολωνία. Η κυρία Σαργκεντίνη για τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, συνάδελφο ε, για το Σολντανόσκ ε, 1989 νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ελπιδοφόρο συμβάν και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αλλά και για εμάς εδώ στη Δύση. Ένα πολύ ελπιδοφόρο λοιπόν συμβάν ε, το οποίο ε, προωθεί και προάγει το κράτος δικαίου ε, και την θετική αλλαγή. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ απολύτως με την ανάλυση που κάνατε για την κατάσταση στην Πολωνία και θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό. Η άρνηση ε, μιας δικαστικής απόφασης ε, για ε, την υλοτόμηση σε ένα δάσος είναι ένα πραγματικά άνευ προηγουμένου γεγονός. όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με το προσφυγικό ζήτημα. Η απειλή προς έναν δημοσιογράφο για τη φυλάκισή του για ένα βιβλίο που, με το οποίο δεν συμφωνεί ένας υπουργός. Όλα αυτά είναι πολύ ανησυχητικά. Το ερώτημα είναι κατά πόσο πρόκειται για συστηματική ε, παραβίαση του κράτους δικαίου. Εγώ μπορώ να πω ότι έτσι φαίνεται. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε κατά πόσο αρκεί ένας απλός διάλογος και αν υπάρχει τέτοιος διάλογος. Γιατί είναι αμφίδρομη αυτή η διαδικασία όλες οι δικές μας επιθυμίες ε, και όλες μας οι ελπίδες ε, για διάλογο από τη δική μας πλευρά δίνουν περισσότερο ε, δικαίωμα στην πολωνική κυβέρνηση να προχωρήσει δικέ της νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς δεν έχετε βάλει όλα τα χαρτιά στο τραπέζι. Όμως νομίζω ότι έχουμε σιγά σιγά περάσει από το στάδιο του διαλόγου και πρέπει ε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε πια το χρόνο, γιατί η Βαρσοβία ε, αξιοποιεί ασφαλμένα ε, και καταχράτα αυτού του χρόνου. Ευχαριστώ κυρία Βίνμπεργκ για το EFDD. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πολλά ακούσαμε σήμερα εδώ. Και πρέπει να πω, μα πού πηγαίνουμε πού πάει ο κόσμος. Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να είναι εύλογες, αλλά από εκεί μέχρι να πούμε ότι ασκούμε τέτοιου είδους πίεση στην Πολωνία, δεν ξέρω. Τα πολωνικά προβλήματα θα πρέπει να το λύσουν οι Πολωνοί στην Πολωνία. Κάπου θα πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή. Εγώ νομίζω ότι υπερβάλλουμε. Συμφωνώ με άλλους ομιλητές από την Πολωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Ο πρώτος αντιπρόεδρος λέει ότι ε, εφόσον όλοι τηρείτε το χρονικό όριο, μπορεί να ακούσει όλες τις παρεμβάσεις σας και να απαντήσει συνολικά. Παρακαλώ, λοιπόν, ζητώ την επιθαρχία σας. Παρακαλώ, Βάρβαρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν έχουν όλοι επίγνωση το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2005 αποφάσισε ότι 1η Αυγούστου είναι η μέρα αλληλεγγύης και ελευθερίας, ακριβώς για ε, να μνημονεύσουμε την ε, συμβολή της ε, Πολωνίας ε, στη δημοκρατία και την ελευθερία. Είναι μια σημαντική ημέρα, όχι μόνο για την Πολωνία, αλλά και για την Ευρώπη. Και το φετινό καλοκαίρι έχει αποδείξει ότι και ο δικός μας λαός ε, θέλει να είναι ελεύθερος. Η στήριξη προς ευρωπαϊκές αξίες ε, ε, συνεχίζει ακάθεκτη. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους σε 150 πόλεις στην Ευρώπη για να περασπιστούν την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δεν ήταν εκεί για τα εργασιακά, για τις συντάξεις και το καθεξής. Όλοι όσοι κατέβηκαν στο δρόμο το έκαναν για να διαμαρτυρηθούν κατά των αλλαγών στην πολωνική δημοκρατία. Δεν θέλουμε να είναι προσχηματική η δημοκρατία στην Πολωνία. Δυστυχώς όμως η πολωνική κυβέρνηση δεν υπαναχωρεί ε, και δεν ε, προτείνει επικοδομητικές λύσεις για την αποκατάσταση της κατάστασης. Και μάλιστα οι υπουργοί απέριψαν ε, πρόσκλησή σας προς τις Βρυξέλλες για να έρθουν να τα συζητήσετε όλα αυτά από κοινού. Μήπως θεωρείτε ότι η Ρώσκα ακριβώς επειδή ήταν δική του ιδέα ε, αυτή η δικαστική μεταρρύθμιση, ότι θεωρείτε ότι δεν κατανοεί λοιπόν την ε, σοβαρότητα και τη βαρύτητα της κατάστασης σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρείτε ότι κατανοεί τι συμβαίνει. Ίσως θα ήταν καλύτερο να τον συναντήσετε κατά πρόσωπο, ε, γιατί θα έχετε τις καλύτερη εικόνα της κυβέρνησης. Κύριος ε, I will speak Polish. Θα μιλήσω και εγώ πολωνικά. Την ώρα που εορτάζουμε την επέτειο των γεγονότων του 1980, του Αυγούστου 1980, τώρα όμως η ίδια η πολωνική κυβέρνηση είναι και είναι και τον πρόεδρο Βαλένσα. Αυτό που κάνει η σημερινή πολωνική κυβέρνηση είναι να καταστρέφει την ελευθερία και την αλληλεγγύη και να υπονομεύει τα θεμέλια της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς για την υπομονή σας απέναντι στην πολωνική κυβέρνηση και για την αντικειμενική σας εκτίμηση και αξιολόγηση του συστημικού κινδύνου σε βάρος του κράτους δικαίου. Και δεν είστε μόνος σα κύριε Τίμερμας, εσεί και το Κολέγιο των Επιτρόπων. Εκατομμύρια Πολωνών συμμερίζονται τις ανησυχίες σας. Και οι δεκάδε χιλιάδες διαδηλωτών του Ιουλίου και αυτοί εκφράζουν τις ίδιες ανησυχίες. Και πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν για να υποστηρίξουν, να υπερασπιστούν το Σύνταγμα και την ανεξαρτησία των δικαστών και σε μεγάλες πόλεις, αλλά και σε δεκάδες μικρές πόλεις. Ερώτηση. Πώς θα προχωρήσετε εν ώψη των πολωνικών απαντήσεων για, και εν ώψη του όσα, των όσων έγιναν ήδη το 2015 όταν το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάσισε να μειώσει τη δική του ανεξαρτησία και σε σχέση με το άρθρο 7 και υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης των ε, αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου σε μια χώρα μέλος. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει το βήμα να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για διαδικασία επί παραβιάση έχοντας υπόψη και το τι συμβαίνει με τον οργανισμό των ε, τακτικών δικαστηρίων. Οι άνθρωποι στην, ε, στις διαδηλώσεις φώναξαν ότι δεν υπάρχει ελευθερία χωρίς αλληλεγγύη και βεβαίως και χωρίς ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Λόπεθ Αγγιλάρ, δύο λεπτά παρακαλώ, τηρήστε όλη τον χρόνο των δύο λεπτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, στα αγγλικά, τώρα στα ισπανικά. Πολύ Είπαμε από το 2008 ότι η κρίση δεν είναι χρηματοπιστωτική αλλά πολιτική αξιών και αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού προγράμματος. Υπάρχει ένας ε, εθνικισμός ο οποίος αναδύεται σε ορισμένες περιπτώσεις αφορά συγκεκριμένα εκλογικά συστήματα όπως το πολωνικό. Πολλές φορές ε, ακούσαμε τις δύο αντιρρήσεις ε, going political, σαν να μην ήταν το κράτος ε, δικαίου ένα πολιτικό ζήτημα. Και δεύτερον είναι η υποκριτική θυματοποίηση, λες και υπήρχαν δύο μέτρα και δύο σταθμά μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής της Βενετίας και αυτό αφορά και άλλους ανεξάρτητους ε, δικαιοδοτικούς μηχανισμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το ΕΔΑΔ. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι προωθούν τη δημοκρατία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την άρνηση της συνταγματικής δημοκρατίας. Κύριε Τίμερμανς, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σας ακολουθήσουμε μέχρι τέλους. Άρθρο 7. Η διαδικασία επιπαραβάση. Και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολη η εκκίνηση αυτής της διαδικασίας γιατί χρειάζεται συμφωνία του Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει θα σας ε, ακολουθήσουμε και αυτό δεν αφορά μόνο τη διαδικασία επιπαραβάση αλλά και την ε, κινητοποίηση, τη χρήση του άρθρου 7. Γιατί μιλάμε για ε, παλινοδίες και αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις. Δυστυχώς η Πολωνία είναι ένα ιδιαίτερα λυπηρό παράδειγμα. Η κυρία Βίκστρεμ. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς για τις άοκνες προσπάθειές σας να βρείτε μία λύση. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη απόλυτα, με απόλυτη σαφήνεια ότι η πολωνική κυβέρνηση στην ουσία κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να καταρρύψει κάθε μορφή ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Τη στιγμή που η κυβέρνηση άρχισε αυτή την αποδόμηση, τη στιγμή που αμφισβητούνται και ανθρώπινα δικαιώματα, ανατρέχω στη, ε, ε στη λογοτεχνία. Τι είχε πει ο Γκόμπροβιτς δεν δέχομαι τα δόγματα, οι ιδεολογίες ή θεσμούς. Θα πρέπει να σταθώ στα πόδια μου. Αλλά δυστυχώς ήμουν Πολωνός, διακατέχομαι από πολωνικότητα και έπρεπε να ζήσω στην Πολωνία. Τη στιγμή που δεν ήμουν πλέον Πολωνός, αλλά μόνο άνθρωπος. Θα πρέπει να ανατρέξουμε σε αυτές τις σκέψεις ε, βλέποντας αυτή την κατάσταση. Δεν μιλάμε για ε, Πολωνία, αλλά για ανθρώπινη υπόσταση. Και αυτό θα πρέπει να είναι και το μήνυμα προς την κυβέρνηση. Δηλαδή, εκεί που απέτυχαν θα διατρανώσουμε τη θέλησή μας εμείς. Ο κύριος Σέντο. Για μένα, Κλώτη, το ενδιαφέρον μου φαίνεται ότι είναι ότι οι Ευρωπαίοι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ε, σταθερή, σταθερό, ε, σεβασμό, σταθερό σεβασμό, ξαναλέω, για την ε, αλληλεγγύη και τον ιστορικό της ηγέτη, που δεν φαίνεται να έχει πολωνική κυβέρνηση. Οι πολωνικές αρχές της σήμερον αμφισβητούν την νομιμότητα και αυτών που αμφισβητούν τις πράξεις τους. Η πολωνική κυβέρνηση στηρίζεται στο 37% του 50% που ψήφισαν. Το 1 έκτο δηλαδή των πολωνών ψηφοφόρων. Και δεν νομίζω ότι η πρόθεση αυτών των πολωνών ψηφοφόρων ήταν να καταστήσουν ομήρους τα υπόλοιπα 5 έκτα. Κύριε Αντιπρόεδρε, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι το ίδιο που έβλεπα να έρχεται από την αρχή. Το ίδιο με την Ουγγαρία. Με μία εξαίρεση και με μία μεγάλη διαφορά. Οι, Ουγ, Ούγγροι τουλάχιστον παριστάνουν ότι συνδιαλέγονται μαζί μας όταν τους επισημάναμε ότι ανάβουν κάποια κόκκινα φώτα. Η πολωνική κυβέρνηση ως τώρα δείχνει απόλυτη αδιαφορία. Η πολωνική κυβέρνηση ως τώρα δείχνει αδιαφορία. Και το πρόβλημα είναι ότι πώς θα γίνει διάλογος. Νομίζω ότι έχουμε ευλόγως εξαντλήσει κάθε δυνατότητα διαλόγου. Αυτό σημαίνει ότι ένα πράγμα μόνο μένει. Γνωρίζω πόσο δύσκολη είναι η εφαρμογή του άρθρου 7. Αν όμως παραλείψουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το τελευταίο μέσον που έχουμε στη διάθεσή μας, νομίζω ότι μπορούμε μια χαρά και να παρετηθούμε από από οποιαδήποτε συζήτηση με Πολωνού, Ούγγρου, οποιουσδήποτε, διότι δεν θα μας θεωρούν πλέον σοβαρού. Και για να μας θεωρήσουν σοβαρού, αυτό μα αφήνει μονάχα μια δυνατότητα. Ενεργοποιήστε το αυτά, ενεργοποιήστε το και εμείς θα σας υποστηρίξουμε. Είμαι βέβαιος ότι ο Αντιπρόεδρος θα απαντήσει στο συγκεκριμένο σας σχόλιο. ο κ. Βάιντενχολτσερ. Βρίσκω αξιοπρόσεκτη την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία έρεται στο ύψος του ρόλου της του θεματοφύλακα των συνθήκων. Πολύ θετικό αυτό. Βλέπω μια ξεκάθαρη αντικειμενική στάση. Η πολωνική κυβέρνηση δυστυχώς φαίνεται να ζει σε ένα παράλληλο κόσμο, τον οποίο έχει φτιάξει μόνη της. και κινείται μέσα σε μια ομίχλη ιστορίας, έθνους, αλλά δεν είναι τα ίδια πράγματα οι διαδηλωτέ οι οποίοι κατεβαίνουν κάθε εβδομάδα στους δρόμους. Είναι λυπηρό ότι έχει κανείς μια... Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή έχουν μια απόλυτα διαφορετική αντίληψη από αυτά που συζητούμε. Κάθε χώρα μέλος αποτελεί, συναποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Υπάρχει ένα κοινό κοινοτικό και κτημένο και τα κριτήρια της Κοπενχάγης ίσχυσαν για όλες τις χώρες οι οποίες συζήτησαν να ενταχθούν και τελικώς εντάχθηκαν. Δεν μπορούμε λοιπόν να είμαστε αδιάφοροι για το τι συμβαίνει στην Πολωνία. Η Πολωνία είναι ένα σημαντικό συστατικό μέρος της Ευρώπης. Θα έλεγα μάλιστα ότι χωρίς Πολωνία η Ευρώπη θα ήταν ένας ε, ακέφαλος κορμός. Είναι σημαντικό αυτό να ακουστεί ως μήνυμα και από, τα, από τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στους δρόμους. Στηρίζω επίσης την θέση να προσπαθήσουμε να συνομιλήσουμε με την πολωνική κυβέρνηση. Η πρόσκληση που απίφθινε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν είναι σημαντική και θεμελιώδης. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις όπου κάποιος αρνείται να συμμετάσχει στο διάλογο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιο σημείο και πρέπει να πούμε δηλαδή πού βρίσκεται το σημείο της μη επιστροφής. Και εγώ νομίζω ότι το σημείο αυτό σιγά σιγά το προσεγγίζουμε. Θα πρέπει λοιπόν τότε να βγάλουμε το χαρτί του άρθρου 7 και διότι οφείλουμε να έχουμε πώς και τι μπορεί να συμβεί άλλο και από άλλες και σε άλλες χώρες μέλη. Ο κ. Ζεντόφσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς για την εμπλοκή σας. Ε, θαυμάσια η ομιλία σας και δεν το λέω διότι είμαστε φίλοι το λέω όμως διότι έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τα λόγια σας, αλλά και για την κατανόηση που δείχνετε του προβλήματος και της νοοτροπίας των Πολωνών. Από τη δική μου σκοπιά είναι σημαντικό να ειδούμε, εγώ ήμουν πολύ δυσαρεστημένος με την κατάσταση στην Πολωνία που είδα φέτος το καλοκαίρι. Βλέπω ότι πράγματι η πολωνική κυβέρνηση Είμαι υπερηφάνος που η πολιτική κυβέρνηση συναποτελεί μέρος του μέρους, του, ε, της ομάδας Βίσεγκρατ. Θα μπορούσα να είμαι ικανοποιημένος. Δεν είμαι όμως. Επαναλαμβάνω και έχω πει πολλές φορές ήδη ότι ήμουν αντίθετος με οποιαδήποτε κύρωση κατά της πολωνικής κυβερνήσεως. Τώρα όμως, όταν μιλούμε για την Σολινταρνόσκ και το 1980, θα επαναλάβω τα λόγια του Πολωνού συναδέλφου μου εγώ έρχομαι από τη Τσεχοσλοβακία και είναι διαφορετική η δική μας εμπειρία από, την, από της Πολωνίας. Όμως στις 23 Αυγούστου του 1968 οι Πολωνοί στρατιώτες σκότωσαν ανθρώπους στην Τσεχία, στην Τσεχοσλοβακία τότε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορώ να εορτάσω την... Μάλλον μπορώ να εορτάσω την επέτειο 1980, όχι όμως το 1968. Διότι εάν χάσουμε τις δημοκρατικές αρχές, εάν χάσουμε τη δυνατότητα διαλόγου, θα καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου η πολωνική κυβέρνηση θα εγκαταλείψει πλέον τις αρχές της δημοκρατίας. Κύριε Γκυγιώμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς αγαπητέ κύριε Τίμερ μας για την δράση που έχετε αναλάβει, την αποφασιστική δράση με σεβασμό των αρχών της Ένωσης μέσα σε όλη την περιπλοκότητά τους και βεβαίως και με τα εργαλεία που διαθέτουμε. Συμφωνώ με πολλές από τις ε, ανησυχίες και ερωτήσεις που εκφράστηκαν και για την συνέχεια των γεγονότων και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η δημοκρατία στην Πολωνία. Θα ήθελα και εγώ το δικό μου μήνυμα να είναι σαφές. Το Κοινοβούλιο αγωνίζεται υπέρ του κράτους δικαίου. Έχω μια ερώτηση τώρα, κάπως γενική. Προμηνών μετέβη στην Πολωνία και άκουσα με ιδιαίτερη ευαισθησία τα λόγια των Πολωνών της κοινωνίας των πολιτών. Τα όσα εξέφρασαν για τη δημοκρατία, για την προσήλωσή τους στις ευρωπαϊκές ιδέες. Και είδα ότι υπήρχε και σημαντική κινητοποίηση προς την Ευρώπη. Πέραν των νομικών εργαλείων που διαθέτουμε και της ενδεχόμενης χρήσης τους, ποια είναι η δική σας αίσθηση σχετικά με την προσήλωση των Πολωνών στις ευρωπαϊκές ιδέες και ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα θέλατε να τους απευθύνετε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ιντφέλτ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Επίτροπο Χαίρομαι για τα λόγια του και θα χαιρόμουν ακόμη περισσότερο να δω και δράσεις που να οδηγούν στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία, διότι οφείλουμε να αναλάβουμε δράση όχι μόνο για να εξασφαλίσουμε την ισχύ του κράτους δικαίου σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για να δείξουμε και κάποια ε, στάση απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Βεβαίω και έχει αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα γράφει το άρθρο 2 τη συνθήκη, που ε, με τη θέλησή της ε, προσυπέγραψε η πολωνική κυβέρνηση, η Πολωνία. Και είναι και το πρώτο άρθρο ουσία στη συνθήκη. Όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν. Νομίζω ότι δεν πρόκειται μόνο για την άσκηση, την επιβολή των όρων της συνθήκης, πρόκειται και για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του πολωνικού λαού, του οποίου τα δικαιώματα παραβιάζονται και δεν είναι θέματα μονάχα δικαιοσύνης. Μιλήσατε πριν και για την υλοτόμηση του δάσους και για τα δικαιώματα των προσφύγων, αλλά και τα δικαιώματα των γυναικών, του συνέρχεστε, της ελευθερίας του τύπου, των μη κυβερνητικών οργανώσεων των πανεπιστημίων. Πρόκειται για παραβιάσεις συστηματικού χαρακτήρα. Δύο τελευταία σχόλια. Αναμένουμε και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την ενεργοποίηση του άρθρου 7. Όμως θα πρέπει και εμείς να λάβουμε τις δικές μας ευθύνες και να εγκρίνουμε σχετικό ψήφισμα. Δεύτερο, η δημιουργία του μηχανισμού του άρθρου 7 ήταν αποτέλεσμα της άρσης στην ηγεσία της Αυστρίας του Γιώζεφ Χάιντερ. Ο μηχανισμός λοιπόν αυτός που πρότεινε το Κοινοβούλιο οφείλει να ισχύει απέναντι σε όλες τις χώρες μέλη με ισότιμο τρόπο. Και ελπίζω ότι σε αυτό θα μας υποστηρίξετε όπως θα υποστηρίξουμε και εμείς εσάς, η κυρία Γκόμες. Προέρχομαι από μία χώρα, την Πορτογαλία, η οποία δεν παραβίασε το κράτος δικαίου και απειλήθηκε με οικονομικά μέτρα γιατί δεν ανταποκρίθηκε σε δεκαδικά στοιχεία ενός κανονισμού και προτάθηκαν τέτοιες, τέτοια επώδυνα μέτρα κατά της Πορτογαλίας. Στην Πολωνία μιλάμε για παραβίαση του κράτους δικαίου κατά σοβαρότατους τρόπους, ιδιαίτερα ως προς την ανεξαρτησία του συστήματος της δικαιοσύνης και ως προς τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, δικαιώματα των προσφύγων και ούτω καθεξής και Τίποτα δεν θα είχε γίνει κατά της Πολωνίας αν δεν είχαμε αντιδράσει κατά της Ουγγαρίας που επίσης παραβίασε κατάφορα το κράτος δικαίου. Υποστηρίζω την Επιτροπή που αντιδρά άμεσα. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 7, αλλά θα πρέπει να είναι θαραλέα η Επιτροπή και να δράσει και με την ε, παρακράτηση των πόρων από το κοινωνικό ταμείο. Αν λοιπόν δεν τηρείται το γράμμα του κράτους δικαίου, τότε τα διαρθρωτικά ε, κονδύλια θα πρέπει να αποσύρθουν μέχρι ότου αποκατασταθεί η νομιμότητα. Θα υποστηρίξουμε την Επιτροπή σε αυτή τη την προσπάθεια, διότι δεν πρόκειται μόνο για την Πολωνία, αλλά για το κράτος δικαίου και βασικά θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους άνδρες και γυναίκες που αντέδρασαν ε, μέσα στα πλαίσια της επανάστασης του Γκτάνσκ. Ο κύριος ε, Γέσεκ. Θα ήθελα να απαντήσω στους συναδέλφους που μίλησαν για υπερβολική πίεση κατά της Πολωνίας. Βεβαίως η Πολωνία είναι ε, μέλος της συνθήκης της Λισαβόνας και αν δεν τηρείται το γράμμα της συνθήκης, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει και αυτό κάνει επιτελεί το καθήκον της ε, και φυσικά δεν μας, ε, κατασ... Ε, δεν μας καθιστά ευτυχής το ότι αντιδρούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι πολωνικό μόνο το θέμα, διότι υπάρχουν κοινέ αξίες και κανόνες και όπως είπε ο πρώτος αντιπρόεδρος, τα πολωνικά δικαστήρια ασχολούνται με θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγοράς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα τα δικαστήρια. Φοβάμαι όμως ότι υπάρχει και ένα σοβαρότερο θέμα γιατί η πολωνική κυβέρνηση δεν θέλει να ξεκινήσει ένα διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πέρα από τις επίσημες λοιπόν διαδικασίες, θα ήθελα να κάνω έκκληση σε όλους έτσι ώστε να έρθουμε σε επαφή με τους Πολωνούς ομολόγους και να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα κατά κάποιο τρόπο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε και από τη δική μου πλευρά σας ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς για το όσα έχετε πράξει εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τώρα. Εγώ συγχαίρω και πάλι τον πολωνικό λαό όπως έπραξαν και άλλοι για την θαραλέα εξέγερση του 1980 και τότε έγινε γνωστό για όλους, σε όλους μάλλον το όνομα Σολινταρνόσκ που ενέπνευσε ελπίδα σε όλες και όλους μας και αυτό το πνεύμα ελευθερίας, ανεξαρτησίας, ανεξαρτησίας του τύπου και της δικαιοσύνης είναι κάτι που τότε δεν υπήρχε αναγκαία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Όμως πάλι τώρα τίθεται θέμα ελευθερίας και δικαιωμάτων και τα πολλά εκατομμύρια Πολωνών, ανδρών και γυναικών που βγήκαν στους δρόμους φέτος το καλοκαίρι ζητούν και αυτοί τώρα την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Διότι βρίσκονται σε κίνδυνο οι πολωνικές και οι ευρωπαϊκές αξίες και αρχές. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, κέριο θέμα. Και κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα ακόμα πιο ξεκάθαρα λόγια από μέρους σας. Πρόκειται για συστηματική παραβίαση του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών. Η πολωνική κυβέρνηση, διευκρινίζω, δεν είναι το ίδιο με την Πολωνία, καταστρέφει, υπονομεύει την διάκριση των εξουσιών, χωρί την οποία ε, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ελευθερία και ούτε βεβαίως ελευθερία στην ενιαία αγορά. Η ανεξαρτησία και η ελευθερία του τύπου, τα δικαιώματα των γυναικών, ακόμα και το περιβάλλον, η προστασία του δάσου του Μπιέλοβιτ, Παρόλε τι σχετικέ αποφάσει. παραβιάζεται. Κύριε Αντιπρόεδρε, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξεκινήσει την ενεργοποίηση του μηχανισμού του άρθρου 7, τότε υπονομεύει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εσωτερικά αλλά και απέναντι στις γειτονικές μας χώρες οι οποίες αναμένουν από εμάς να δείξουμε στεναρή στάση σε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι και εσείς κύριε Τίμερμανς είπατε ότι πολιτικά είμαστε ουδέτεροι όταν πρόκειται για κράτος δικαίου. Ποιος σας πιστέψει όμω εν ώψη των προσφάτων εξελίξεων, μιλήστε καθαρά, Πετε καθαρά τι θέλετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς συγκεκριμένα επηρεάζετε την κοινή γνώμη στην Πολωνία υποστηρίζοντας την αντιπολίτευση. Και έτσι τάσεστε αντίθετη με την εκφρασμένη θέληση του πολωνικού λαού. Δεν είχα την εντύπωση ότι ήταν παράνομη ή αντιδημοκρατική η εκλογή που εξέλιξε την παρούσα πολωνική κυβέρνηση, γίνονται ελεύθερε δημοκρατικές εκλογές και εκεί κατεβαίνουν οι υποψήφοι όπως επιθυμούν. Πέστε λοιπόν καθαρά περί τίνο πρόκειται, μιλήστε καθαρά, διότι εγώ θεωρώ ότι αυτό που θέλετε εσείς είναι μονοκαλλιέργεια. Θέλετε να καταστρέψετε τις εθνικές χώρες και στην περίπτωση της Πολωνίας αυτό σας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρουν τα δάση που θα κοπούν, σας ενδιαφέρει μονάχα ότι η Πολωνία ασκεί μια μεταναστευτική πολιτική που δεν ταιριάζει στις ιδέες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε και σε κάποιους άλλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δηλαδή, δεν κάνουν τα πράγματα όπως θα ήθελατε εσείς. Α, όμως υπάρχουν ελεύθερες χώρες στην Ευρώπη, κυρίαρχες, οι οποίες σέβονται και υπερασπίζονται την εκφρασμένη θέληση των λαών. Αυτό σημαίνει στην Πολωνία. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα υποστηρίξω διαδικασία παραβίασης κατά της πολωνικής κυβέρνησης. Αντίθεση με τη χώρα μου, τη Γερμανία, η Πολωνία είναι ελεύθερη χώρα, κυρίαρχη, η οποία αποφασίζει μόνη της για το μέλλον του λαού της πάντα είναι θετικό να ακούμε απόψεις από όλο το πολιτικό φάσμα. Από την αρχή άκουσα ότι, είπα μάλλον, ότι υπό τον κορώνα 206 θα ακούσουμε και μέλη εκτός της Επιτροπής μας. Αλλά για να γίνει αυτό και να έχουμε και αρκετό χρόνο για τον πρώτο αντιπρόεδρο να απαντήσει, θα ήθελα να παρακαλέσω τα μη μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ να μην υπερβούν το ένα λεπτό. Ιδάλλως ε, θα καθυστερήσουμε και δεν θα έχουμε χρόνο για την απάντηση του πρώτου αντιπροέδρου. Παρακαλώ λοιπόν να μείνετε στο ένα λεπτό. Ο κύριος Αρνέκη πρώτος, παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω το εξής. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε απάντηση ε, προς τους Πολωνούς δικαστές είπε ότι αρνείται να επέμβει σε εσωτερικά ζητήματα της πολωνικής δικαιοσύνης. Τώρα όμως τι κάνατε ακριβώς αυτό. Αυτό δεν είναι λοιπόν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σε πολλές ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούνται εδώ και από συναδέλφους που πήραν το λόγο προηγουμένως, ε, εφαρμόζονται αντίστοιχες και ταυτόσιμες λύσεις με αυτές που προωθεί αυτή τη στιγμή η πολωνική κυβέρνηση. Και τέλος, έχω την εντύπωση ότι σε αυτή την αίθουσα ε, δεν επιχειρηματολογεί κανείς, ε, εσείς μάλλον, με γεγονότα και στοιχεία, αλλά με μύθους σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Πολωνία. Και κλείνοντας, δεν νομίζω ότι μιλάτε για το κράτος δικαίου στην Πολωνία. Περισσότερο έχει να κάνει με το γεγονό ότι δεν θέλουμε να δεχθούμε του μετανάστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ποιε είναι οι προσδοκίε αυτή τη στιγμή στην Πολωνία. Σαφώ εργασία και καλή μισθή, δικαιοσύνη και ασφάλεια και το 80% των ε, Πολωνών γνωρίζουν ότι η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν μια ε, καλή και αξιοπρεπή ζωή. Η κυβέρνησή μας θέλει να ακολουθήσει την οδό της ε, σύγκρουσης και εγώ θα ήθελα να τονίσω την ανεξαρτησία μας εξαιτίας της συμβολής μας ε, στην διαδικασία της μεταμόρφωσης στην Ένωση και στον κόσμο. Θα ήθελα η Πολωνία να είναι ένας αξιοσέβαστος εταίρος. Είμαι πεπισμένος ότι πρέπει να ε, σεβαστούμε την εξουσία των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, να θυμάστε ότι και η συνθήκη της Λισαβόνας κυρώθηκε και υπεγράφει από την ε, κυβέρνηση αυτή κατά την προηγούμενη θητεία της. Και τώρα για τις κυρώσεις. Δεν είναι το ένα έκτο το οποίο θα πληγεί από τις κυρώσεις. Είναι τα υπόλοιπα πέντε έκτα που θέλουν να είναι στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η Πολωνία είναι μια χώρα που βασίζεται στο κράτος δικαίου, είναι μια δημοκρατική και φιλοευρωπαϊκή χώρα και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί προσπαθείτε να αντιστρέψετε ε, αυτόν τον ε, φιλοευρωπαϊκό χαρακτήρα της Πολωνίας. Μιλήσατε για τις κοινέ μας αρχές. Αλλά τι αρχές έχουμε τελικά εδώ ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασιστήκαμε στις χριστιανικές αρχές και αξίες. Και μα θυμίζετε τώρα αυτό που ε, είχε πει ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο ότι η Ευρώπη χρειάζεται την Πολωνία. Μιλάτε για αλληλεγγύη. Να σα υπενθυμίσω λοιπόν, ε, Επίτροπε, ότι το Ε, ή μάλλον η αλληλεγγύη στην Πολωνία έχει φταφτεί κάτω από το Nord Stream. Τελικά δεν υπάρχει καμία αλληλεγγύη. Ε, το σημερινό σύστημα ε, ήταν ιδιαίτερα ισχυρό εναντί των αδυνάμων. Αυτή, αυτός είναι ο λόγος. Στη Βαρσοβία υπήρχαν άνθρωποι που τους πέταξαν έξω από τα σπίτια τους γιατί κυβερνούσε ε, η πολιτική πλατφόρμα. Και πώς είχε κατάσταση με τα παιδιά στη Γερμανία, στο Jungen Ans. Η Επιτροπή είχε πει ότι δεν ήταν δική της αρμοδιότητα να επερασπιστεί αυτά τα παιδιά. Λέτε λοιπόν ότι ουσιαστικά υποστηρίζετε τους σοσιαλιστές και τους ε, λαϊκιστές. Συνάδελφοι, μέχρι τώρα υπήρχε πειθαρχία. Ας συνεχίσουμε έτσι. Ε, δέχτηκα να ακούσουμε τους επόμενους ομιλητές πέραν τη επιτροπή με τον κανόνα, με, τον, με την προπόθεση να μιλήσετε για ένα λεπτό. Εάν δεν το τηρήσετε όμω, θα σταματήσει εδώ η συζήτηση. Ο κύριος Κάρσκι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να αφορά την αλήθεια. Γι' αυτό δεν κατανοώ την ομιλία του κυρίου Τίμερμανς. Αν θέλετε να μιλήσετε για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε το εξής. Ε, δεν υπάρχει ε, λύση που να μην ισχύει στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, εμείς προβάλαμε λύσεις που έχουν εισαχθεί και ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και εσείς λέτε ότι ότι δεν θέλετε οι Πολωνοί δικαστές να λαμβάνουν τηλεφωνήματα από το κόμμα. Ίσως θα πρέπει να το συζητήσετε με τον κύριο Τούσκ και να σας μιλήσει τι συνέβαινε όταν ήταν εκείνος πρωθυπουργός, γιατί τότε ένας δημοσιογράφος κάλεσε έναν δικαστή από την πόλη που καταγόταν ο Τούσκ και είπε ότι θα ήθελε να υπάρχει μια συγκεκριμένη σύνθεση του δικαστηρίου για μια υπόθεση και αυτός ο άνθρωπος ακόμα κατέχει τη θέση του. Έγκελ. Θα αντιταχθώ προσπαθώ να ε, συνεχίσετε αυτή η συζήτηση από μέλη που δεν προέρχονται από την ε, Επιτροπή μας και γίνεται ένα ιδιωτικό κατηγορητήριο εδώ. Συμφωνώ μαζί σας. Πέντε ομιλητές έλαβαν το λόγο χωρίς να ανήκουν στην Επιτροπή μας και νομίζω ότι αρκεί αυτό Ήμασταν αρκετά ευέλικτοι δυνάμει του άρθρου 206. Δεν μπορώ να λάβω το λόγο. Με συγχωρείτε πολύ, με συγχωρείτε πολύ. Εάν ακούσατε αυτά που μόλις προείπα, μίλησαν πέντε μέλη που δεν προέρχονται από την Επιτροπή. Γι' αυτό θα ήθελα ο πρώτος αντιπρόεδρος να απαντήσει στους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ακούσατε τι είπα. Θα ακούσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο, τις απαντήσεις του. Παρακαλώ, ησυχία. Δεν δέχομαι διαδικαστικό. Προχωρήστε κύριε ε, Αντιπρόεδρε. Δεν ε, δέχομαι αυτά που είπε ο κύριος Φρανκ Έγκελ. Δεν κατανοώ γιατί δεν μας δώσατε το λόγο. Κύριε Τιούρεκ, ισχύει ο το άρθρο 206. Σας παρακαλώ να σταματήσετε. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήμουν φοιτητή το 80 και θυμάμαι πολύ καθαρά το ότι ε, είδα τον Λέχ Βαλέσα που μίλησε για τις κοινέ ευρωπαϊκές αξίες. Ε, ήμουν φοιτητής και μετά στρατιώτης και θυμάμαι πολύ καλά ότι το όραμα της Ευρώπης φαινόταν αιώνιο. Ότι δεν θα υπήρχε αποδόμηση, ότι χρειαζόμασταν σταθερότητα. Και η, η μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ε, κράτησε την Ευρώπη αδιέρετη. Θα μπορούσε βεβαίως να παραμείνει έτσι κατά διαφορετικό τρόπο, γιατί ανεξάρτητα με το ποιος είναι επικεφαλής στη ε, ε, Ρωσία σήμερα ή χτες ήθελαν μια διαιρεμένη Ευρώπη και την θέλουν διαιρεμένη και στο μέλλον. Μαχόμαστε για την ευρωπαϊκή ενότητα με βάση κοινές αξίες, με βάση το κράτος δικαίου και το νόμο και την τήρηση του νόμου της συνθήκης των συνθήκων που έχουν κυρωθεί από κυρίαρχα κοινοβούλια. Και αν στις συνθήκες αυτές είναι χρέος της Επιτροπής να διασφαλίσει την τήρησή τους που κύρωσαν, η ίδια η Επιτροπή θα αναλάβει αυτό το καθήκον σοβαρά αν και πολιτικά μπορεί να είναι επώδυνο. Θεωρώ ότι η Πολωνία σήμερα είναι πιο κυρίαρχη, ελεύθερη, έχει πιο ασφαλή σύνορα από ό,τι είχε κατά πολλούς αιώνες του παρελθόντος. Για χίλια χρόνια η Πολωνοί πλέον είναι πιο ελεύθερη μετά από χίλια χρόνια για να αποφασίσει για το μέλλον της. Εάν η Γερμανία ήταν πιο δυνατή θα είχε 300 χιλιόμετρα σύνορα λιγότερα πιο προς τα μέσα και το ίδιο ίσχυε και για την πρώην Σοβιετική Ένωση θα είχε καταστρατηγήσει τα σύνορά της κατά 300 χιλιόμετρα εξανατολών. Μιλάμε λοιπόν για, μια, για ένα κυρίαρχο κράτος, για την Πολωνία, έναν εξάρτητο κράτος που δεν ίσχυε για εκατοντάδες χρόνια. Και δεν μπορώ προσωπικά να φανταστώ μία επιτυχή Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς μία Πολωνία που να ευημερεί. Γιατί μιλάμε για την ε, ημαρμένη της Ευρώπης όταν μιλάμε για μία Πολωνία που ευημερεί. Τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Και αυτοί που λένε ότι η Επιτροπή δεν τα βλέπει σωστά. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε την ίδια άποψη με την Επιτροπή της Βενετίασης. Της Βενετίας, η οποία προέβη στην ανάλυση μετά από αίτημα της πολωνικής κυβέρνησης. Άρα η πολωνική κυβέρνηση ζήτησε αυτή την ανάλυση. Όταν την έλαβα όμως και δεν της άρεσε, αποφάσισε να την αγνοήσει. Αν λέτε λοιπόν ότι η Επιτροπή δεν κατανοεί τα πράγματα, σας παρακαλώ να ξέρετε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτή μας την εκτίμηση. Όταν συζητήσαμε το ζήτημα στο Συμβούλιο το Μάιο, αυτό πολλές φορές το παραβλέπουμε, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία υποστήριξε τη θέση της Επιτροπής. Άρα η Επιτροπή δεν δραμώνει της και το Κοινοβούλιο επίσης αντέδρασε, δηλαδή και τα τρία θεσμικά όργανα κάνουν ό,τι μπορούν για να επιληθεί αυτό το ζήτημα στην Πολωνία. Είχαμε τις απαντήσεις της πολωνικής κυβέρνησης και θα απαντήσουμε. Αλλά ως προς τα θέματα που εφήγησαν σήμερα. Μην δεχτείτε την άποψη ότι άλλα κράτη έχουν παρόμοιες λύσεις. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει ένα κράτος όπου ο υπουργό Δικαιοσύνης μπορεί να απολύσει αυθαίρετα έναν δικαστή, να τον απολύσει, να προσλάβει άλλους. Δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα αλλού. Κάθε φορά που τίθενται ζητήματα επιτάπητος και κάποιος φωνασκεί «Μα δεν ισχύει κάτι τέτοιο», δείτε, δείτε τα κείμενα Αυτή είναι η ουσία. Εμείς στείλαμε συστάσεις που είναι λεπτομεριακές. Η πολωνική κυβέρνηση μας έστειλε δύο επιστολές ζητώντας ε, αποσαφηνήσεις. Εμείς τις δώσαμε και άρα ας παραμείνουμε στα κείμενα. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον ή κάπως ηρωνικό είναι αυτό το συνεχές αίτημα για τήρηση του γράμματος του νόμου και σεβασμού, ο οποίος δεν είναι όμως αμφίδρομος. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Εμείς θέλουμε τον διάλογο Όποιος θέλει μπορεί να μου κάνει προσωπικές επιθέσεις, να λέει ότι είμαι γελίος, αναξιοπρεπής, ό,τι θέλει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να συνεχίσουμε αυτή την πορεία διαλόγου. Κάποια στιγμή θα πρέπει να προβούμε σε επιλογές θα παρετηθούμε του ζητήματος γιατί δημιουργεί πολιτικές δυσχέρειες ή θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα διφορούμενο. Δεν θα παρετηθούμε επειδή υπάρχουν πολιτικές δυσκολίες, διότι οι συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι πολύ σοβαρές όταν μιλάμε για διαχωρισμό των εξουσιών και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας όταν δεν τηρείται ο διαχωρισμός των εξουσιών. Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής σε αυτό. Δεν μιλάμε μόνο για το κράτος δικαίου, αλλά την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις, τις πτυχές όλα εξαρτώνται από την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και από τον ε, διαχωρισμό των εξουσιών. Εάν αυτό αμφισβητηθεί, θα πρέπει να αντιδράσουμε και να μην επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι ο πυρήνας του ζητήματος. Γιατί στο κάτω-κάτω, οι μόνοι που θα προσδιορίσουν την τύχη της Πολωνίας είναι οι ίδιοι οι Πολωνοί. Όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε όταν δεν τηρείται το γράμμα των συνθήκων που έχουν κυρώσει κράτη-μέλη, τότε θα πρέπει να αντιδράσουμε και να το στυλιτεύσουμε γιατί διαφορετικά θα απεκδιόμασταν των ευθυνών μας. Θα πρέπει να το κάνω και εγώ και η Επιτροπή. Και για να είμαστε σαφείς, γιατί υπάρχει έλλειψη σαφήνειας, το θέμα δεν είναι προσωπικό. Εγώ μιλώ εξ ονόματος της Επιτροπής και η Επιτροπή είναι ενωμένη επί του θέματος και μιλώ εξ ονόματος και της συλλογιστικής πολλών κρατών μελών. Αφού σας άκουσα, έχω την εντύπωση ότι μιλώ και εξ ονόματος της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ο Πρόεδρος Μωράης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρώτη Αντιπρόεδρε. θα συζητήσουμε το θέμα και μεταξύ των συντονιστών. Σας ευχαριστώ για τα εισαγωγικά σας σχόλια καθώς και για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη και προχωρούμε με την ημερησία διάταξή μας. Um, Ο πρόεδρος, εφόσον αποχωρείτε παρακαλώ πράξετε το σε ησυχία. Χωρίς ε, φασαρία γιατί έχουμε και άλλα θέματα στην ημερησία διάταξη. Κύριε Τζούρεκ, παρακαλώ ένα λεπτό για το διαδικαστικό σας θέμα. Ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν αμφισβητώ το δικαίωμά σας να περιορίσετε τον κατάλογο των ε, μελών που θα μιλήσουν και που δεν είναι τακτικά μέλη της Επιτροπής. Είπατε όμως ότι θα επιτρέψετε σε όλους να λάβουν το λόγο όσοι επιθυμούν. Ο καθηγητής ο Κρασνοτάρσκι ζήτησε να λάβει το λόγο ήδη από την αρχή και τελικώς δεν του δόθηκε. Εγώ ζήτησα το λόγο με τον ίδιο τρόπο όπως ο Φρανκ Έγγελ σας παρακαλώ, και πάλι μου το δώσετε, σας παρακαλώ να τηρείτε όμως ίση μεταχείριση. Σα, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που θέτετε το διαδικαστικό σας θέμα με ήρεμο τρόπο. Έδωσα το λόγο σε πέντε βουλευτές μη μέλη της ε, Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών. Νομίζω ότι ήταν λογικό αυτό και έτσι επέτρεψα και στον ε, Αντιπρόεδρο να μπορέσει να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πάντως για το δικαστικό σας θέμα. Νομίζω ότι φάνηκα όσο ήταν δυνατόν ε, γενναιόδωρος. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Στρατηγική και το ψηφιακό εμπόριο. Εάν είστε έτοιμοι... Το Δεκέμβριο αποφάσισε η Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών να συντάξει γνωμοδότηση για θέματα που το των αρμοδιοτήτων της, ενώ επί της ουσίας αρμοδία είναι η Επιτροπή Ίντα με εισηγήτρια την κυρία Σχάκε. Θα γίνει ή έγινε και η ενδέκατη σύνοδος των Υπουργών του ΠΟΕ και θα δώσω λοιπόν τώρα τον λόγο στην κυρία Μλίναρ για να μπορέσει να τοποθετηθεί σχετικά με το σχέδιο ομοδοτησιός της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε μετά από την θερμή συζήτηση που προηγήθηκε. Ερχόμαστε πλέον πάλι στα συνήθη θέματα της ημερησίας διατάξεως. Το ζήτημά μας που είναι το ψηφιακό εμπόριο και διαμεθοριακές συναλλαγές και που είναι ε, καθημερινά πράγματα για όλων των ειδών και μεγεθών τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πράγματα που δεν υπήρχαν πριν από 15 χρόνια καθόλου. Όμως τώρα είναι σημαντική η επιρροή τους στην αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των χωρών μελών. Αυτή, ωστόσο, η αλλαγή ε, μεταμορφώνει και το εμπόριο όπως το γνωρίζαμε. Κάποτε μιλούσαμε μονάχα για τη ροή αγαθών. Τώρα όμως οι υπηρεσίε που είναι το 3, τα τρία τέταρτα της ευρωπαϊκής οικονομίας ε, μπορούν και παρέχονται και διαμεθοριακά. Οι εγχώριες νομοθεσίε ε, διαμορφώνουν την ψηφιακή οικονομία. Οι δε σχετικέ συμφωνίες θα πρέπει να παρακολουθούν τον ρυθμό αυτό. Όμως δεν συμβαίνει αυτό και αυτό αποτελεί πρόκληση για μας. Την Ευρωπαϊκή δηλαδή Ένωση ως κοινότητα αξιών αλλά αποτελεί και μεγάλη ευκαιρία για να άρουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο τα διεθνή πρότυπα. Με σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής σφαίρας που μέχρι τώρα αποκλείονταν από τις, ευρωπαϊκές, από τις ε, διεθνείς συμφωνίες. Το κεκτημένο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα επιτρέπει και την ελεύθερη διακίνηση των δεδομένων. Χρειάζεται όμως να λαμβάνεται υπόψη για τις αποφάσεις των ε, τρίτων χωρών και να κωδικοποιηθεί ένας από τους μηχανισμούς για τις μεταφορές δεδομένων και προτείνονται εκεί και διάφορες δυνατότητες και επιλογές. Λαμβάνονται νέες μορφές μιας ψηφιακής τελειοθυρίας. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι νέοι κανόνες για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων μπορεί να εμποδίζουν την διαχείριση δεδομένων σε τρίτες χώρες εάν αυτές δεν ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δηλαδή. Με λίγα λόγια και για να ολοκληρώσω, η προώθηση υψηλών προτύπων για την μεταφορά δεδομένων και η υψηλή τους προστασία θα πρέπει να συμβαδίζουν. απευθύνω στον επόπτη προσωπικών δεδομένων δύο ερωτήσεις και ζητώ απάντηση προς όφελος όλων μας. Πρώτο, κατά την άποψή σας, ποιο είναι το υψηλότερο επίπεδο δυνατό σε διεθνείς συμφωνίες για την προστασία των δεδομένων και δεύτερο, ποιες ρήτρες υπάρχουν ήδη συμφωνίες για την ροή των προσωπικών δεδομένων και για τον χειρισμό τους. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας καθώς και για, την, ε, για το σχέδιό σας, ε, Αγγέλικα. Έχουμε και ορισμένους κοιόδης εισηγητές. Α, εσείς είστε, μάλιστα, αντικαθιστάτε τον κύριο Ράντε, κυρία Μεζόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον Μιλιράντε που δεν μπορούσε να εδώ σήμερα. Σκιώδης εισηγητής θεωρεί ότι το διαδίκτυο, νέες τεχνολογίες και ψηφιοποίηση επηρεάζουν κάθε πτυχή τη καθημερινότητάς μας από τον ε, τρόπο ε, που λειτουργούμε στην καθημερινή μας ζωή μέχρι και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχουν ε, αυξηθεί κατακόρυφα οι ροέ δεδομένων τα τελευταία χρόνια με μια τεράστια οικονομική συμβολή στην παγκόσμια ανάπτυξη οι εμπορικέ ε, ροέ δεδομένων συνεχώ αυξάνονται ακόμα και παρά την κρίση. Παρ' όλα αυτά, πολλοί ε, υφιστάμενοι κανόνε δεν ε, ανταποκρίνονται σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Πολλέ χώρε χρησιμοποιούν μέτρα προστατευτισμού για να πάρουν ένα θέμητο πλονέκτημα ή για άλλου λόγους και αυτό αποβαίνει σε βάρος των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ε, η ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί ότι η ε, ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και το ίσο πεδίο ανταγωνισμού είναι απαραίτητες σημασία σε στοιχεία για την ενιαία αγορά. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε και την επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ παράλληλα βέβαια σεβόμαστε πλήρως και την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κανόνες που να ανταποκρίνονται στις ε, διεθνείς εξελίξεις, ε, προσδιορίζοντας ε, μια ευρωπαϊκή θέση που να καλύπτει αυτές τις προϋποθέσεις για την οικοδόμηση περαιτέρω εμπιστοσύνης, αμοιβές εμπιστοσύνης και με χώρες. Θα πρέπει η Επιτροπή να συνεχίσει τις συζητήσεις με διεθνείς εταίρους για πιθανές αποφάσεις επάρκειας. Τέλος, ο Σκιώδη θεωρεί και ελπίζει ότι θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προσβλέψει συνέχιση τη συνεργασία με την εισηγήτρια και τους υπόλοιπου Σκιώδη για να το πετύχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Κραπίνη είναι η Σκιώδης από πλευρά του Χελστών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα Νομίζω ότι καλώς ε, εκφέρει γνώμη για αυτό το θέμα η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Μιλήσαμε πολύ για τις συνθήκες σήμερα το πρωί, επομένως αν δείτε τις συνθήκες βλέπετε ότι πέραν της ε, υπεράσπισης ε, των, αξιών, ευρωπαϊκών αξιών και τη αναπτυξιακή βοήθεια προ αναπτυσσόμενε χώρε, θα πρέπει να καλύψουμε και να προάγουμε και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα και τις πολιτικές ελευθερίες και δικαιώματα. Επομένω είναι ευπρόσδεκτη η γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι όλες ε, οι εμπορικές ε, συμβάσεις και η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικά ισχυρό όπλο για την προάσπιση των αξιών μας σε αυτές τις χώρες, αρκεί να πρόκειται για ίσα ε, πρότυπα και να μην ε, και δίκαια πρότυπα και να μην ε, πλήττουν τους εταίρους μας ή κάποιον από τους εταίρους. Θα πρέπει να υπάρχουν τέτοια πρότυπα για την, για την επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί τέτοια στοιχεία μπορεί να βρει κανείς σε εμπορικές πολιτικές πίεση που ασκείται στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η έκθεση της πρωτοβουλία πρέπει να έχει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα. Ελπίζω έτσι να γίνει και με τη δική μας συμβολή. Η ψηφιακή επανάσταση έχει ε, Μα έχει φέρει αντιμέτωπο με νέα ζητήματα σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην Ευρώπη και διεθνώ. Νομίζω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών να ε, γίνονται σεβαστά. Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το καθεξής. Όλοι λοιπόν ε, δεχόμαστε ερωτήσεις από τις εκλογικές μας περιφέρειες σε ό,τι αφορά το σύστημα που έχουμε εγκαθιδρύσει για την προστασία δεδομένων. Θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες ε, ηλεκτρονικού εμπορίου και διασυνοριακών ροών δεδομένων προκειμένου να ε, προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Βέβαια δεν μπορούμε να πάμε προς τα πίσω, πρέπει να αναπτύξουμε ε, το ε, ηλεκτρονικό και το διασυνοριακό εμπόριο. Παράλληλα όμως θα πρέπει να έχουμε και ένα σύστημα προστασίας. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εταίροι μας ακολουθούν τους ίδιους κανόνες και προϋποθέσεις με εμάς. Μίλησα και για την ε, ΣΥΤΑ και για την ΤΙΤΙΠ και για κάθε άλλη μεγάλη ε, εμπορική συμφωνία την οποία διαπραγματευόμαστε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να αξιοποιούμε αυτές τις εμπορικές συμφωνίες, παράλληλα όμως να υπάρχουν ε, πολύ συγκεκριμένα εχέγγυα κατά πρακτικών ντάμπινγκ και του ανταγωνισμού γιατί υπάρχει ακόμα αυτό το πρόβλημα. Άλλο πρόβλημα είναι βέβαια η διαφθορά, ιδίω στις φτωχότερες χώρες. Νομίζω ότι τελικά οι εμπορικέ συμφωνίε μπορούν να αξιοποιηθούν για την καταπολέμηση και τη φτώχεια και τη διαφθορά. Γι' αυτό μαζί και με την ομάδα των σοσιαλιστών προσπαθούμε να συμβάλλουμε ε, και να στείλουμε μια παρέμβαση για αυτή την έκθεση. Ελπίζω να υπάρχει καλή συνεργασία για αυτή την έκθεση. Κύριε Στόλτον, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και του Χιώδη για τα όσα έχουν κάνει μέχρι τώρα. Ε, μιλώ με πολλές ιδιώτε, γιατί είμαι και εισηγητή για την γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΙΜΚΟ για τους καταναλωτές. Όμως θα προσπαθήσω να ε, μείνω μόνο στα της ε, ΛΥΜΠΕ. Από πλευρά ΕΣΥΑΡ ε, χαιρετίζουμε του ε, στόχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διευκόλυνση του ηλεκτρονικού εμπορίου και τα όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι τεράστιε τομέ ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερο εξαγωγέα τέτοιων ε, υπηρεσιών. Θα πρέπει λοιπόν όμω να ενεργούμε προδραστικά για να ενθαρρύνουμε ακριβώ το θεμητό ανταγωνισμό στη νέα αυτή ψηφιακή εποχή. Γιατί το εμπόριο μα βοηθά και μα ευνοεί όλου και την Ευρώπη και τι ε, υπόλοιπε χώρε. Πρέπει όμω να τα κάνουμε όλα σωστά. Το βασικό είναι να δούμε πώ θα διασφαλίσουμε την προστασία των ε, κανόνων προστασία δεδομένων σε όλο τον κόσμο, αλλά να μην παρεμποδίζεται και η ελεύθερη ροή δεδομένων. Δεν μπορούμε να αποδυναμώσουμε του κανόνε μα για την ε, ψηφιακή προστασία και δεν προτείνει κανεί κάτι τέτοιο. Όμω θα πρέπει να διασφαλίζεται και η ελεύθερη ροή δεδομένων. Αυτό είναι ο πιο σημαντικό παράγοντα για την διασφάλιση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ψηφιακού εμπορίου και όλοι ε, μου προτείνουν ότι οι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών δεν είναι ο καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα και τα θέματα ε, συμφωνιών επάρκεια, γιατί δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε μια τέτοια συμφωνία μετά από τρία χρόνια, για παράδειγμα, αν έχει αλλάξει κάτι σε μία από τι δύο χώρε εταίρου. Γι' αυτό και εμεί στο ECR θεωρούμε ότι ε, εδώ ο καλύτερο τρόπο θα ήταν συγκεκριμένε συμφωνίε επάρκεια όπως αυτή που ε, διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, συνάπτει τέτοιες συμφωνίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα είναι καλό και για την Επιτροπή Λίμπε. Ιδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος, η προστασία δεδομένων ε, να αξιοποιείται ως ένα έμεσος τρόπος για να παρεμποδίζεται το εμπόριο ως ε, μη δεσμολογικό εμπόδιο. Δεν θέλουμε λοιπόν να δούμε κάτι τέτοιο. Υπάρχει όμως ε, τρόπος, πιστεύω, ήδη ε, αξιοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στηρίζουμε λοιπόν την Κομισιόν στα όσα κάνει και περιμένουμε με υπομονησία να δούμε και την έκθεση και να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους κοιότες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Όλμπρεχτ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συνεχίζοντας με τα όσα υπόθηκαν προηγουμένω για την προστασία δεδομένων και για το θέμα του ψηφιακού εμπορίου, πρέπει να θεσπίσουμε ορισμένες βασικές αρχές για τον κλάδο και επειδή δεν πρόκειται μόνο για διμερείς εμπορικές συμφωνίες, αλλά και έχουμε και την ε, διυπουργική ε, του ΠΟΕ στα τέλη της χρονιάς. Εκεί θα εξεταστούν όλα αυτά τα ζητήματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει θέση για βουλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δούμε πώς μπορούμε ε, να τα εξετάσουμε όλα αυτά εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων. Γιατί βέβαια υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Ιδίως για παράδειγμα, για το θέμα της προστασίας δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφύσεως έχει διαφορετική στάση από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση η προστασία δεδομένων είναι ε, θεμελιώδης δικαίωμα. Γι' αυτό και συμφωνώ και με τον κύριο Ντάλτον ότι για εμάς δεν θα ήταν σωστό να θέσουμε την προστασία δεδομένων σε ε, εμπορικές συμφωνίες, γιατί είναι θεμελιώδης δικαίωμα. Δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευση. Όμω, άλλε τρίτε χώρε μπορούν να ανέρχονται στο δικό μα επίπεδο προστασία. Να μην το βλέπουμε λοιπόν ω θέμα ελευθέρω συναλλαγών, αλλά να λέμε ότι μπορούν να υπάρξουν τέτοιε συναλλαγέ γιατί υπάρχουν κοινά πρότυπα. Γι' αυτό μετά τα ψηφίσματα που υιοθετήσαμε για τις διαπραγματεύσεις ε, TTIP και TISA εδώ στην Επιτροπή μας, είπαμε ότι οι συμφωνίες επάρκειας θα πρέπει να είναι η πρώτη απόπειρα, αυτή είναι η προτεραιότητα δηλαδή, και αν δεν επιτυχάνονται τότε ε, το... η δεύτερη επιλογή στα εμπορικά ζητήματα είναι να υπάρχει πάντα μια οριζόντια ρήτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων που ε, δεν ε, αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευση, δεν ε, εμπίπτει σε αιρεσιμότητε. Ισχύει πάντα. Πρέπει να δούμε αντίστοιχε διατάξει στι χώρε εταίρου και βέβαια ε, υπό τους κανόνες GATT αυτά τα πρότυπα, όπως για παράδειγμα στην προστασία δεδομένων, θα πρέπει να αξιοποιούνται για Άλλου ε, σκοπού. Δεν θα πρέπει μάλλον να αξιοποιούνται για άλλου σκοπού. δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει πρόθεση πέραν τη προστασία δεδομένων, σε όλε τι περιπτώσει όπου δεν υπάρχει συμφωνία επάρκεια για την προστασία δεδομένων, να υπάρχει λοιπόν μια αυτόνομη οριζόντια ρήτρα ε, για να διασφαλίζεται η προστασία δεδομένων. Δεν νομίζω ότι είναι ακαθόδε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει ευρεία συνένεση. Έχουμε ψηφίσματα. Είναι σημαντικό όμω να το λέμε ξανά και ξανά για να είναι σαφή και η θέση μας προ τους ε, εμπορικούς εταίρους μας και να κατανοούν ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα για μας. Ευχαριστώ Γιάννη. Η κυρία Γκόμες παρακαλώ. Κοιτάξτε, να μην είμαστε αφελεί και να θεωρούμε ότι οτιδήποτε σχέση με το εμπόριο είναι μια χαρά. Εξαρτάται αν είναι δίκαιο εμπόριο. Διότι αν δεν είναι δίκαιο θα κάνει πλουσιότερους τους πλούσιους και ισχυρούς και θα φτωχύνει του υπόλοιπου. Και αυτό βλέπουμε τώρα. Α σταματήσουμε αυτές τις ανοησίες ότι δήθεν ότι η σχέση με το εμπόριο είναι θαυμάσιο. Δεν είναι. Και ο, ο δικός μας ρόλος είναι να το κάνουμε δίκαιο, ρυθμίζοντά το, για όλους. Και βεβαίω και εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άποψη αυτή, συμφωνώ ότι η προστασία προσωπικών δεδομένων είναι και θεμελιώδες δικαίωμα, αλλά και θεμελιώδες στοιχείο για την ασφάλεια των συναλλαγών. Αν θέλουμε να προωθήσουμε το εμπόριο, πρέπει να προωθήσουμε και την προστασία των δεδομένων. Αλλιώς δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη στις εμπορικές συναλλαγές. Πάρα πολύ λοιπόν κρίσιμο στοιχείο και βεβαίως και ανθρώπινο δικαίωμα και θεμελιώδες δικαίωμα, όπως είναι και για μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που όμως δεν συμβαίνει για άλλους και ιδιαίτερα εννοώ τους Αμερικανούς εταίρους μας. Η ερώτηση που έχω ωστόσο απευθύνεται τον εισηγητή και στην Κομισιόν. Και έχει ως εξής. Μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλούμε για διευκόλυνση του ψηφιακού εμπορίου που είναι όλο και περισσότερο το εμπόριο που βλέπουμε πια στην εποχή μας εάν αγνοούμε όπως εξακολουθούμε να αγνοούμε τους κινδύνους του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος που διευκολύνει το ψηφιακό εμπόριο εάν ε, αγνοούμε επίσης τον ε, ε, κίνδυνο φοροδιαφυγής. Κινδύνους που ανοίγει το ψηφιακό εμπόριο αν δεν υπάρχουν κανονισμοί και ρήτρες. Για παράδειγμα αυτό το εικονικό νόμισμα bitcoin τώρα με την Εστονική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιοι φαίνεται είναι πολύ ευχαριστημένοι που λένε ότι η Εστονία ξεκινά, ε, εισάγει ένα ε, εικονικό νόμισμα. Μα αυτό είναι απλούστατα ένα εργαλείο για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, για την εξαπάτηση μέσω θογοροδιαφυγής των κρατών μας και ούτω καθεξής. Εμείς τι κάνουμε μέσα σε όλα αυτά μπορούμε να συνεχίσουμε, να, συνεχίσουμε να αγνοούμε τις εξελίξεις αυτές εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί σε ό,τι αφορά την διευκόλυνση του ψηφιακού εμπορίου και του εμπορίου γενικότερα, αλλά με δίκαιο τρόπο. Ευχαριστώ, Άννα. Έχουμε όμως στις 11 η ώρα ψηφοφορία. επιστρέφω λοιπόν τον λόγο στην Αγγέλικα. αφού πρώτα ακούσουμε όμως τον κύριο Μεν από την ETPS. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την πρώτη σας ερώτηση. Η προστασία δεδομένων και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να προστατεύονται καλύτερα και μέσα στις διεθνές, διεθνείς ε, συμφωνίες. Τα είπε αυτά και ο Πρόεδρος Γιούνκερ στην ομιλία του State of the Union. Είπε τότε ότι η προστασία δεδομένων είναι θεμελιώδης δικαίωμα και η προστασία που θα ενταχθεί σε εμπορικές συμφωνίες για εμάς χρειάζεται μια οριζόντια ρήτρα που να προβλέπει ότι γίνονται απολύτως σεβαστές οι διατάξεις αυτές. Είμαστε σύμφωνοι με αποφάσεις adequacy decisions, όπου η TPS έχει συμβουλευτικό ρόλο. Αυτή είναι η απάντησή μας στην πρώτη σας ερώτηση. Για τη δεύτερη ερώτηση, ε, είμαστε δηλαδή η υπόπτηση για, τα, για των ε, προσωπικών δεδομένων. Η DPS δεν ζητεί τη γνώμη της όσον, όσον δεν υπάρχει επιρροή για τα προσωπικά δεδομένα. Όταν υπάρχει τότε είναι αρμόδια η αρχή μας. από την αρχή της διαπραγματευτικής εντολής, δηλαδή όπως γίνεται και με τη Γενική Διεύθυνση σωστερικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου η αρχή μας σεβάστηκε απολύτως τη διαδικασία εγγράφων περιορισμένης χρήσεως. Ωστόσο, η DPS για την διαπραγματευτική εντολή για τις εμπορικές συμφωνίες δεν έχει ζητηθεί η γνώμη της. Τον Φεβρουάριο του 2010 η αρχή μας εξέδωσε γνωμοδότηση για δική της πρωτοβουλία, μάλλον με δική της πρωτοβουλία, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων άκτα για το άρθρο 41 παράγραφος 2 του κανονισμού μας, σύμφωνα δηλαδή με το άρθρο αυτό. Το 2012, όταν δημοσιεύθηκε στον τύπο το κείμενο της Συμφωνίας Άκτα, ζητήθηκε τότε από την αρχή μας, ε, μάλλον η, αρχή μας εξέδωσε δεύτερη γνωμοδότηση με δική της πρωτοβουλία. Ο επισήμως δεν έχει ζητηθεί τώρα η γνώμη της ETPS. Ε, μόνο ανεπίσημα και μόνο επειδή μια χώρα μέλος μας ειδοποίησε, είμαστε εν γνώση του εγγράφου. Θα είναι καλή ιδέα λοιπόν οι συνομοθέτες να ενισχύσουν τον ρόλο του EDPS όταν θα συζητούνται θέματα διεθνών συμφωνιών που έχουν επιρροή στα προσωπικά δεδομένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε ήδη διεξαγάγει μια συνάντηση των ενδιαφερομένων μερών. Έχουμε κάποια θέματα ακόμη ανοιχτά. Όπως είπαν και οι συναδελφοί μου, έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το Κοινοβούλιο να αποκτήσει μια στέρεα θέση που να ενισχύεται από σημαντική πλειοψηφία και να μένουμε βεβαίω στη συνεργασία με τους κοιόδης συζήτητες. Ε, ευχαριστώ. Η συζήτηση του σχεδίου θα γίνει στις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 28 θα πρέπει να έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες και στις 23 Νοεμβρίου θα γίνει ψηφοφορία. Θα κάνουμε την ψηφοφορία στις 11 η ώρα, άρα να διακόψουμε για 10 λεπτά και να επανέλθουμε στις 11 και παρακαλείστε όλοι να έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες έτοιμες.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 Mr. Chairman, can we get on with this, please? μπορούμε να προχωρήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως και θα προχωρήσουμε, απαντά ο Πρόεδρος Μωράες. Όταν θα καθίσουν όλες και όλοι οι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ, καθίστε για να μπορέσουμε να αρχίσουμε με την ψηφοφορία. Καλά λοιπόν. Αρχίζουμε. Έχω δύο εκθέσεις του κ. Γέσεκ. Πρώτα για τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οικονομικό έτος 2018. Νομίζω ότι είστε όλοι σε ρυθμό ακόμα καλοκαιριού και γίνονται πολλές ιδιωτικές συζητήσεις αλλά είμαστε έτοιμοι, είστε και εσείς έτοιμοι. Καλά λοιπόν, ε, γνωρίζω ότι ορισμένοι επίγεστε να αρχίσουμε, ας αρχίσουμε λοιπόν. Ε, έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2018 με εισηγητή τον κύριο Γέσικ. Παράγραφος 1, συμβαστική 1, αρχίζει η ψηφοφορία. Ελπίζω ότι δεν έχετε ξεχάσει πώς ψηφίζετε. Πατήστε το πράσινο κουμπάκι. Λέει ο πρόεδρος. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2α αρχίζει. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 2β. Συμβαστική 2β αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Η... Μα αρχίζει η ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος. Τέλος. Απερίφθη. Τροπολογία 12, τμήμα 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τροπολογία 12, τμήμα 1. Πέρας. απερίφθει 12, τμήμα 2. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 15 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 αρχίζει. Τέλος. Εγκρίνεται. 18 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. απεριφθεί. Συμβαστική 3. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30. Όχι, λέει ο πρόεδρος, με συγχωρείτε. Λάθος. Μια στιγμή σας παρακαλώ. Τροπολογία 26. Έναρξη. 26. Πέρας. Απορρίπτεται. 27. Ε, έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 28. Έναρξη. Πέρας. απορρίπτεται 29 έναρξη πέρας απορρίπτεται 30 έναρξη πέρας απορρίπτεται 31 έναρξη πέρας Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 39. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 40. Πέρας. Απερίφθη. 41. Πέρας. Εγκρίνεται. 42. Έναρξη. Πέρας. Απορρίπτεται. 43 έναρξη. Πέρασε. Απορρίπτεται. 44 έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. 45 τμήμα πρώτο. Όχι. Τμήμα δεύτερο, λέει ο πρόεδρος. Α, πρώτο τμήμα. Ζητώ και πάλι συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 45 τμήμα πρώτο. Έναρξη ψηφοφορία. Τμήμα πρώτο. Ένα. Πολλά λάθη κάνω σήμερα, λέει ο πρόεδρος. Πέρας. Απορρίπτεται. 45 τμήμα δεύτερο. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 45 τμήμα τρίτο. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Έναρξη. Πέρας. εγκρίνεται. 48 τμήμα πρώτο. Πέρας. Εγκρίνεται. 48 τμήμα δεύτερο. Πέρας. Εγκρίνεται. Η ψήφος τώρα για το τροποποιημένο κείμενο αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται με 40 ψήφους υπέρ, 9 κατά και καμία αποχή. Και ερχόμαστε στην τελευταία ψηφοφορία που είναι πάλι του κυρίου ε, Γέσεκ για τον προϋπολογισμό του 2018. Πρόκειται για τροπολογίες επί του προϋπολογισμού αρχίζει για την ΔΥΜΠΕ 6024. 6024. Επιγράφεται, αυτό ψηφίζουμε, επιγράφεται ΛΥΜΠΕ 6024. Πέρας, εγκρίνεται. Λίμπε 6021 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Ελίμπε 6001 μάλλον. 6001. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 6002. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.003 υπέρ. Μάλλον έναρξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.012 έναρξη. Πέρας. Απερίφθη.

Πέρας. Εγκρίνεται. 6.026. Έναρξη. απεριφθη 60-32. 6.032. Έναρξη. Πέρας. Απερίφθη. 6034 έναρξη. Πέρας. Απερίφθη. 6037 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 6033 έναρξη. Πέρας. Απερίφθη. 6.043 έναρξη. Πέρας. Απερίφθη. 6.045 Πέρας. Απερίφθη. 6.018 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.047 έναρξη. Ψηφοφορίες. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτή. 6.025 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.027. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.030. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Έναρξη. πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.020 έναρξη. Α, συγγνώμη συνάδελφοι. 6.035 πρώτα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 6.020 έναρξη ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 6.004 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 6.005 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.006. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.007. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.014. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.008 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.022 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.009 έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.010. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.029. Έναρξη. Πέρας. Εγκρίνεται.

και 44 άρχεται πέρας εγκρίνεται 6.046 άρχεται πέρας εγκρίνεται 6046 6.017, 6.051 ταυτόσημες. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.050. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 6.016, 6.049 ταυτόσιμες. Έναρξη. Πέρασε. Εγκρίνεται. Η τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Έναξη ψηφοφορίας. Πέρας. 41 ψήφοι υπέρ, 9 κατά, 0 αποχές, συγχαρητήρια προς τον εισηγητή. Ευχαριστώ συνάδελφοι, εδώ τελειώνουν οι ψηφοφορίες και η συνεδρίαση. Υπάρχει κάτι άλλο από τα διάφορα. Εντάξει, φτάσαμε στο τέλος ε, του καλοκαιριού, αυτό είναι ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ. Επόμενη συνεδρίαση στις 3 ε, το μεσημέρι της 4 Σεπτεμβρίου.